Στο θέμα 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Θέλω να σας υπενθυμίσω σε όλους σας ότι αυτή η συνεδρίαση βρίσκεται, μεταβιβάζεται και στο ε, διαδίκτυο, στο web και θα ήθελα να έχετε και τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για την ψηφοφορία διότι θα προχωρήσουμε όταν θα έρθει η ώρα των ψηφοφοριών και θα χρησιμοποιήσουμε τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013. Ο εισηγητής παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα. Λάβαμε ένα email από την κυρία Τσεσκόβα σχετικά με την τροπολογία 9 και μας είπε ότι θέλει να αποσύρει αυτή τη συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα, αυτό το είχαμε πληροφορηθεί, έχει αποσυρθεί και έτσι νομίζω στη συνέχεια τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε Λοιπόν, ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας, συμβιβαστικής τροπολογίας 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα στη συνέχεια, συμβιβασμός 1 και άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πάλι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και αυτό το τμήμα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 προφορική τροποποίηση από πλευρά του άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, τροπολογία 10, άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 12, άρχεται, πέρας, απορρίφθηκε. Τροπολογία 13, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο συνολικά υπέρ ε, με συγχωρείτε πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ ένας εναντίον δεν είχαμε αποχές εγκρίθηκε Συγχαρητήρια λοιπόν όσον αφορά τον εισηγητή και προχωρούμε στη συνέχεια έχουμε χορήγηση απαλλαγών για τις υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Με την απαλλαγή 2009 για τον... Ο κύριος Σταυρακάκης είναι εισηγητής ε, για τον έλεγχο των οργανισμών. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ψηφίζουμε. Και αρχίζουμε με την προφορική τροπολογία αριθμός 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 5, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Όχι. 7. Η 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Πρώτο τμήμα. Αρχίζει είναι προφορική η τροπολογία, διορθώνεται το πρόεδρος. Αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 29 με μια προφορική τροπολογία. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 23 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 33 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 34 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 36 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 37 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 38 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 39 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 40 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 41 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 42 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 44. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. 47 υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εκτιμώντας F 2 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα ούτως τροποποιημένο αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνονται 24 υπέρ, κανένας κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε τώρα στην απαλλαγή 2009 για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, την ΕΑΑ. Πάντοτε είναι εισηγητής ο κύριος Σταυρακάκης. Λοιπόν, πρόταση απόφασης για την απαλλαγή. Τροπολογία 1 και 2 μαζί. Είναι ίδιες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. Πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 25 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, κανένας κατά. Τελικό ψήφισμα. Παράγραφος 1 της ΛΥΜΠΕ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δύο της ΛΥΜΠΕ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δέκα Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 με μια προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 12, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 13, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας Απορρίπτεται. 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 με μια προφορική τροπολογία αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Λίμπεθ, Προπολογία 8, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Έγκρινεται. 24 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 αρχίζει η ψηφοφορία με την προφορική τροπολογία. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 26 αρχίζει η ψηφοφορία. 26 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 της ΛΥΜΠΕ αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Με προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Πέρας εγκρίνεται 32 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 34 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 35 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 33 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά το ψηφισμό που τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κανένας κατά και μία αποχή.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 την, πρόταση απόφασης για την απαλλαγή στο σύνολό της. Εγώ νομίζω ότι τη σημειώσαμε, την ψηφίσαμε. 25 την υπερψήφισαν, δεν υπήρχε καμία εποχή το ψηφίσαμε έτσι δεν είναι. Δεν ήταν το κλείσιμο των λογαριασμών λέει η γραμματεία. Να το ξαναψηφίσουμε για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Μιλάμε για την πρόταση απόφαση απαλλαγή. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ. Εγώ θυμόμουν ότι το ψηφίσαμε λέει ο πρόεδρος. Να ψηφίσουμε αμπλόκ όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ε, λίστα. Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ λέει ο πρόεδρος. Διότι η συνάδελφος Μακοβέη είναι κατά. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ψηφίζουμε αρχή την πρόταση απόφασης για την απαλλαγή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, κατά και μία αποχή. Πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορια Εγκρίνεται 22 υπέρ, ένας κατά και μία αποχή. Τροπολογία 1 τώρα για το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το γράφει λέει ο Πρόεδρος εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5. Αρχίζει η ψηφοφορία εγκρίνεται 7 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 1 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 2 με μια προφορική τροπολογία αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 6 της ΕΜΒΗ αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ψηφίζουμε συνολικά το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε αρχίζει ψηφοφορία 21 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Πολύ ωραία. Τώρα, ο κύριος Σταυρακάκης θέλει το λόγο. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ο, ο συνάδελφος Σταυρακάκης είναι ο εισηγητής τροπολογίες 1 και 2 στην πρόταση για την απαλλαγή αρχίζει ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 10 όχι καταπέμπτει ψηφίζουμε συνολικά την απόφαση Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Τώρα, πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνολικά την πρόταση όπως τροποποιήθηκε αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Κανένας κατά. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει ζητήσει το λόγο. Dear colleagues, before we vote the resolution, I would like to comment on some of the amendments θα ήθελα πριν ψηφίσουμε να σχολιάσω μερικές τροπολογίες. Αναφέρομαι εδώ στις τροπολογίες που αφορούν στον διαμεσολαβητή για τα φάρμακα και σε εκείνα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για δηλώσεις πάρα πολύ σοβαρές και δεν, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις που τεκπηριώνουν. Το θέμα mediator θα πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς με μια διαδικασία ακριβή και διαφανή. Υπάρχουν άτομα τα οποία πέθαναν και οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να εξετάσουμε ενδελεχώς ε, το θέμα, αλλά όχι σε αυτή την έκθεση περί απαλλαγής. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με την εξειδικευμένη επιτροπή και με μια ακρόαση που θα είναι καλά προετοιμασμένη και όπου θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμενες την περασμένη Πέμπτη. Η διάσκεψη των Προέδρων επέτρεψε μια, μια επίσκεψη ε, και ζήτησε κατεπηγόντως να εξεταστεί το θέμα. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου μπορούμε να δούμε τι δεν πήγε καλά. Θα συμβάλλουμε σε αυτό στην Οριζόντια Επιτροπή. Ε, ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να κάνει εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους για όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Επίσης, ζητούμε ζητήσαμε να γίνει ειδικό λογιστικός έλεγχος για το θέμα αυτό. Εκ μέρου τη πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτές οι τροπολογίε εγκριθούν θα ψηφίσουμε κατά του ψηφίσματος στο σύνολό του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε. Τροπολογία 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 8 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 10 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 11 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 12 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 με προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. 22 δεύτερο τμήμα. Προφορική τροπολογία 22, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται 23 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 24 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Αποσύρθηκε τροπολογία 25. Ναι. Τροπολογία 26. Πέρας. Τροπολογία 27. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 29. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 32. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 33. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άμβη 1. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Η πέντε. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Χέρτζοκ. Ξέχασα την κάρτα μου. Εντάξει. Τροπολογία 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 37 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 40. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 42. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 43. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά το ψήφισμα ούτως τροποποιημένο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ 8 κατά. 9, 9 διορθώνεται ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η κυρία Μακοβέη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. MV4. MV4. Está en V4, En V4, ¿dónde está? Minus, minus. Ok. Passiamo adesso al discarico 2000. Απαλλαγή 2009, Ευρω... Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμου. Ο κύριος Σταυρακάκης είναι πάντα ο εισηγητής και ξεκινάμε με την απόφαση για την απαλλαγή ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 1 μαζί με την τροπολογία 2 που είναι ίδιες και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφασης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ 1 κατά μία αποχή πρόταση για ε, την απόφαση για το κλείσιμο των λογαριασμών ψηφίζουμε την τροπολογική, προφορική τροπολογία 2 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 υπέρ, ένας κατά και μία από εκεί. Τώρα, το ψήφισμα. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 3 και αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συνολικά το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και μία αποχή. Τελευταία ψηφοφορία, πάντοτε είναι η εισηγητής ο συνάδελφος Σταυρακάκης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, δηλαδή για το Frontex. Ψηφίζουμε την απαλλαγή, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 21 υπέρ, ένας κατά μία εποχή για το κλείσιμο των λογαριασμών αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ, έναν κατά και μία αποχή. Ψήφισμα. Τροπολογία λίμπε 1, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. λίμπε Λίμπε 4, αρχίζει ψηφοφορία, προηγούμενη τροπολογία εγκρίθηκε. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Το ψήφισμα αποστροποποιήθηκε, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και μία αποχή. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σέα, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους κοιόδης εισηγητές, τους βοηθούς μου και βεβαίως τη γραμματεία για την συνεργασία την οποία είχαμε κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων μηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την εργασία σας. Γύρισα ακριβώς. Ακριβώς, ναι, <laughs> Δεν ήξερα, του είπα γάλα με καφέ με γάλα. Δεν ήξερα, θυμόμουν. Σε ευχαριστώ. Τι Bene. Passiamo... Τώρα, πάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αριθμός 11 του 2010 η εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης της Γενικής Δημοσιονομικής Στήριξης στις χώρες ΑΚΕ καθώς και στις χώρες Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Ο συνάδελφος Μπέρμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Πρόεδρε, για την εισαγωγή. Να δεσίνα τη μινούτη. Ένα δεκάλεπτο, κύριε. Τότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, συντομότερος από ό,τι προέβλεπα. Λοιπόν, Πρόεδρε, Πρώτα, στον κόσμο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, η υποστήριξη με κονδύλια, η συνδρομή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ήταν απόλυτα υπέρ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπέρ και σε μια ανακοίνωση του 2005 από πλευράς τους μια, στη διακήρυξη των Παρισίων του 2005 οι χορηγοί δεσμευόντουσαν, δεσμεύτηκαν η βοήθεια αυτή να διασφαλίζεται και να παρέχεται μέσω των χωρών και με άμεση υποστήριξη δημοσιονομική. Υπάρχουν δύο μορφές. Η γενική συνδρομή, η δημοσιονομική γενική συνδρομή και εξειδικευμένη, με εξειδικευμένα κονδύλια. Αυτό τώρα οδηγεί στο ότι 48% να είναι το συνολικό ποσοστό αυτής της σύνδρομης όσον αφορά την ευρωπαϊκή ε, συνεργασία για την ανάπτυξη δημοσιονομικά με τη διασφάλιση κονδυλίων. Η υποστήριξη αυτή έχει πολλά προτερήματα. Αυτή είναι η ανάλυση μου. Προτερήματα επειδή όχι μόνο ο μεγαλύτερος όγκος μπορεί να διασφαλιστεί κονδυλίων και υπάρχει και προβλεψιμότητα για σχεδιασμό από την χώρα αποδέκτη. Η χώρα αποδέκτη, η αποδέκτης έχει και μεγαλύτερο, μεγαλύτερη εμπλοκή και μπορεί να εκφράζει και τις επιθυμίες και ανάγκες της. Αυτό εξαρτάται για το πώς η κυβέρνηση σε σχέση με τους χορηγούς μπορεί να συνεργάζεται. Υπάρχουν καλύτερες επαφές δηλαδή. Και ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια εμπλέκονται και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να βελτιώνουν τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή μεγαλύ, υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη από πλευρά τους, μεγαλύτερη εμπλοκή και έτσι έχει θετικό αποτέλεσμα αυτή η σύνδρομη. Ένας διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών χωρών αποδεκτών. Ο πολιτικός αυτός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να υπάρχει ένας καλύτερος εναρμονισμός, ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των χορηγών, ώστε η αποτελεσματικότητα της συνδρομής της βοήθειας αυτής να βελτιώνεται, να αυξάνεται και ένα μεγαλύτερο ποσοστό να μπορεί να διατίθεται. Αυτό είναι η θεωρία βέβαια. Στην πρακτική έχουμε κάποιο, κάπως διαφορετική εικόνα. Έκανε μια μελέτη συνέταξε το ελεγκτικό συνέδριο και εξέτασε και είδε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτούς τους στόχους, πώς τους διατυπώνει, πώς ε, αντιμετωπίζει τους κινδύνους και πώς ε, από την άλλη πλευρά τα προγράμματα συνδρομής τα αναπτύσσει, τα σχεδιάζει και πώς ε, υποβάλλει εκθέσεις ναι, το θέμα είναι για να ε, μπορεί να ε, διαπιστώνεται όχι μόνο αν έχουν διαθεθεί τα χρήματα με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται και αντιμετωπίζει αυτή την ε, συνδρομή για την ανάπτυξη. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει μια ολόκληρη σειρά κριτικών παρατηρήσεων που διαπιστώνει. Έχουν διαπιστωθεί δηλαδή ευάλωτα σημεία, εύτρωτα σημεία όσον αφορά τη μεθοδολογία και τη λειτουργία. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, ίσως θα μπορέσει να τοποθετηθεί στη συνέχεια κιόλας αφορά το, στην έκθεσή του το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκώς ε, εξειδικεύσει τα πράγματα στη στοχοθέτηση για τις επιμέρους χώρες. Είναι δηλαδή υπερβολικά γενικόλογο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την κάλυψη των κινδύνων, δύο κυρίως κινδύνων, να μην καταλήξουν αυτά τα κονδύλια στα χέρια εκείνων που δεν είναι δικαιούχοι και να μπορέσουν τα προγράμματα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Είναι δύο κίνδυνοι που το ελεγκτικό συνέδριο πιστεύει ότι δεν έχουν επαρκώς ληφθεί υπόψη. Και έχουμε και τα προγράμματα τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά, δεν λειτουργούν ε, και δεν σχεδιάστηκαν και δεν λειτουργούν κανονικά ε, αποτελεσματικά όσον αφορά τα αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις δηλαδή δεν είναι ε, δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη σε σχέση με το σχεδιασμό και την κατάρτιση των προγραμμάτων. Γι' αυτό καταλήγει το ελεγκτικό συνέδριο στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε στην έκθεσή της περισσότερο να εδράζεται σε, ε, εδράζεται περισσότερο αυτό είναι η μομφή του ελεγκτικού συνεδρίου σε ενδυνάμει ε, ε ωφελήματα και όχι στα πραγματικά ωφελήματα στο πραγματικό όφελος. Για μας είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το εξής αυτή η ε, δημοσιονομική συνδρομή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μπορεί να είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συνεργασία για την ανάπτυξη. Αν και όταν χρησιμοποιείται σωστά. Χρησιμοποιείται σωστά τι σημαίνει. Σημαίνει τα προτερήματα, τα ωφέλη να μπορούν να απορρέουν όπως τα προανέφερα. Υπάρχει ένα, ένας όρος που είναι του σειρμού και δεν τον, δεν τον βρίσκω αυτό τον όρο ιδιαίτερα θετικό, όμως παρόλα αυτά να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι το mainstreaming, το απέφυγα στην έκθεσή μου το mainstreaming. Είναι του σειρμού αυτός ο όρος το mainstreaming, αλλά όπως και άλλοι όροι, ε, εφόσον χρησιμοποιούνται, ας τους αφήσουμε όσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ως εισηγητή, λοιπόν ανησυχώ ιδιαίτερα με βάση το γεγονό ότι το ελεγκτικό συνέδριο εκπροσωπεί την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει με σύνεση του μεγάλου κινδύνους σε σχέση με τη δημοσιονομική σύνδρομη. Υπάρχει ελλειπή αντιμετώπιση, ελληματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Είτε καταλήγουν αυτά τα κονδύλια σε χέρια μη δικαιούχων, είτε δεν απο... επιτυγχάνεται το ευκταίο αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν σημαντικά να ληφθούν υπόψη είναι αυτά. Μια χώρα λοιπόν που δεν έχει ίσως ένα σωστό λογικό αποτελεσματικό δημοσιονομικό σύστημα αλλά βρίσκεται καθοδόν προς ένα τέτοιο σύστημα μια τέτοια χώρα θα πρέπει να μπορέσει να τύχει μια τέτοια σύνδρομη. Αυτή είναι η σκέψη η οποία βρίσκεται πίσω από αυτή την δυναμική της σε μετεξέλιξη ευρισκόμενης ε, δημοσιονομική ε, σύνδρομη. 12 χώρες ΑΚΕ και 5 χώρες ε, της Λατινικής Αμερικής, 17 χώρες την χάνουν αυτή της δημοσιονομικής σύνδρομης. 17 χώρες βρίσκονται, αυτές οι 17 χώρες πάνω πάνω στον <clears throat> δίκτυο κινδύνου. Αυτό λοιπόν δεν βαίνει καλώς. Πρέπει να έχουμε ένα αυστηρότερο σύστημα monitoring, εποπτείας, να ξέρουμε τι γίνεται με τα κονδύλια σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ελεγκτικό συνέδριο είναι απεσιόδοξο όσον αφορά αυτή την προοπτική. Σε αυτές τις 17 χώρες πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να δούμε τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια. Και αυτό οδηγεί και στην παρατήρηση ότι αν και όταν η δημοσιονομική συνδρομή παρέχεται με αυτόν τον τρόπο, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στις χώρες αποδέκτες ε, που ωφελούνται θα πρέπει να είναι δεδομένος και να λειτουργεί και θα πρέπει να ενισχύεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στις χώρες αυτές. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επενδύσει σε αυτόν τον έλεγχο. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει μια ελληματική κατάσταση σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν θα γνωρίζουν, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν τα αναγκαία στελέχη για να ε, επιτυγχάνεται αυτό ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει και τούτο υπόψη. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει ασκήσει επικρίσεις στο γενικό τμήμα της δημοσιονομικής σύνδρομης. Θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένη λοιπόν η δημοσιονομική σύνδρομη και όχι τόσο γενική στα, στο, στη μορφή και στα πλαίσια της. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά να ενστερνιστούν αυτές τις ιδέες. Η πρόσθετη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ενδυνάμει πολιτικό βάρος και η πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ο πολιτικός διάλογος, διάλογος με τις χώρες αποδέκτες από τις χώρες χορηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικός. Γιατί διαφορετικά αν δεν υπάρχει, αυτός ο, αν δεν υπάρχει αυτή η πολιτική επαφή, τότε κάποια χώρα μπορεί να τύχει συνδρομής, κάποια άλλη όχι. Και θα πρέπει να είμαστε να λειτουργούμε με ενιαία μέτρα και σταθμά, να μην είμαστε ασύνετοι. Η πολιτική πρόσθετη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπονομεύεται. Και εδώ πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα στην δράση μας και θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν αυτή την κριτική, αυτές τις επικρίσεις και να είναι πιο αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη διότι πολλές φορές ακολουθείται μια ξεχωριστή πολιτική από τα κράτη-μέλη χωρίς να υπάρχει συντονισμός των πολιτικών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι λοιπόν σημαντικό να μεριμνήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί όπου υπάρχει εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αντιπροσωπείες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τα αναγκαία στελέχη στη διάθεσή τους, να έχουν την αναγκαία πείρα, την απαιτούμενη πείρα και εμπειρία τα μέλη αυτά, τα στελέχη αυτά για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Αν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη στελέχωση πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν και όσον αφορά τα προσόντα τους και αυτά πρέπει να αναβαθμιστούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση και να έχουμε και μια ετήσια τέτοια έκθεση για την συνδρομή αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Έκενσταν από το Ελεκτικό Συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ στην Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια ε, γενική εικόνα σύντομη σε σχέση με την έκθεση αυτή. Βεβαίω είναι αναπέφευκτο ε, ότι θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα που επεσήμανε ο εισηγητής ε, νομίζω ότι ο συγητής στην έκθεσή του σε αυτό το έγγραφο έκανε, συνόψε πολύ καλά τις δραστηριότητες μας. Όπως ακούσατε από την παρουσίαση, πρόκειται για ένα σημαντικό σκέλος 50% ε, της βοήθειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 50% διοχετεύονται διαμέσου αυτού του μηχανισμού Πρόκειται για χρήματα που δίδονται απευθείας και υπάρχουν ε, πολλές, πολλές δυνατότητες, πολλά δυνητικά πλεονεκτήματα. Αυτό έχει αναγνωριστεί. Γι' αυτό είδαμε ότι είναι η επιλογή που προτιμάται από την διακήρυξη των Παρισίων και από άλλα έγγραφα. Βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό με τρόπο που να είναι προβλέψιμος για τις χώρες αποδέκτριες. Όπως είπε ο κύριος Μπέρμαν, είναι επίσης ένας τρόπος όπου βλέπουμε ότι ε, ε, μπορεί να δημιουργηθεί περισσότερη ιδιοποίηση ευθύνη από τις χώρες αποδέκτες και να βελτιωθεί έτσι η διαχείριση από τις χώρες δικαιούχους. Οι χώρες που λαμβάνουν τα κονδύλια αυτά έχουν, πρέπει παράλληλα να ε, βελτιώσουν τις δημοσιονομικές διαδικασίες, διαδικασίες λογιστικού ελέγχου κλπ Αυξάνεται επίσης το συνέστημα υπευθυνότητας, λογοδοσίας, εμπλέκονται οι χώρες αποδέκτριες με τρόπο τακτικό. Και αυτό γίνεται με έναν διάλογο πολιτικό. Ε, πήγαμε στην Ρουάντα την, το φθινόπωρο και εκεί υπήρχε κάθε μήνα ε, μια συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών των βασικών ε, υπουργείων που ήταν αποδέκτες και των δοτών. Και ε, των χορηγών και είδαμε πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα, τα κονδύλια στα διάφορα υπουργεία. Έτσι βελτιώνεται ο συντονισμός ανάμεσα ε, στους ε, δότες. Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Η Επιτροπή κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσει το σύστημα αυτό, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά αδυναμίες και βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ε, θα αναφερθώ στο θέμα αυτό ε, ε, λεπτομερώς. Θα μπορούσα όμως να πω εκ των προτέρων ότι η Επιτροπή γενικά έχει δεχθεί τα συμπεράσματά μας και η Επιτροπή έχει ένα, μια διαδικασία ευρύτερη με μια πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό που διανεμήθηκε για να ανοίξει ένας ευρύτερος διάλογος και συζήτηση για το θέμα αυτό. Τώρα οι διάφορες παρατηρήσεις. Σε αυτά τα προγράμματα υπάρχουν συνήθως μακρο, ε, στόχοι μακροοικονομικής ε, διαχείρισης ε, και δημοσιονομικής διαχείρισης. Νομίζω ότι είναι παρόμοιοι οι στόχοι στις διάφορες χώρες. Δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ειδικές περιστάσεις στις διάφορες χώρες και ε, επισημάναμε περιπτώσεις όπου οι προτεραιότητες ε, των χωρών έχουν αλλάξει ενώ τα προγράμματα δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχει επίσης τάση, παράσταση στόχοι αυτοί να είναι πολύ γενικοί. Αν πρέπει να είναι χρήσιμοι θα πρέπει να είναι αρκετά σαφείς, αρκετά συγκεκριμένοι, να καταλαβαίνει κανείς τι είναι ακριβώς μια βελτίωση. Αυτό δεν είναι πάντοτε η παράσταση και περίπτωση και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι καταστάσεις για να δούμε τι πρέπει να επιτευχθεί, τι θέλει ο καθένας να επιτύχει. Το δεύτερο μου σημείο έχει να κάνει με, το, με ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η Κομισιόν πρέπει να αναπτύξει και αυτό επίσης αναφέρθηκε από τον εισηγητή ένα σύστημα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων Υπάρχουν μερικοί ειδικοί κίνδυνοι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Ε, δαπανούμε μεγάλα ποσά διαμέσου των κεντρικών κυβερνήσεων, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι που εμπλέκονται σε αυτή όλη τη διαδικασία, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι σε σχέση με την αναπτυξιακή ε, στρατηγική και το ένα πλαίσιο χρειάζεται σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Ε, ο συλλογισμός που ακολουθείται ε, σχετικά με τα ποσά, τα κονδύλια ε, που διοχετεύονται προς κάθε χώρα δεν είναι σαφής. Ε, οι εκταμιεύσεις μπορούν να είναι μάλλον προβλέψιμες. Οι χώρες ξέρουν εκ των προτέρων τι θα λάβουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να κατανοήσει κανείς τα πράγματα με αυτό το υλικό. Γιατί ορισμένες χώρες παίρνουν τόσα πολλά χρήματα και άλλες λιγότερα. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για να μπορέσουν να κρυθούν τα κονδύλια, εκτιμηθούν τα κονδύλια που θα λαμβάνουν οι χώρες. Βεβαίως υπάρχουν εδώ πολιτικά θέματα τα οποία εμπλέκονται. Αλλά δεν ξέρει κανείς που αρχίζει η πολιτική και που λύγει ο συλλογισμός των συμπερασμάτων υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν ένα θεωρητικό πλαίσιο για ε, να αιτιολογούνται οι εκταμιεύσεις και μετά θα προστίθενται οι ε, πολιτικοί παράγοντες. Αλλά θα πρέπει να δούμε απ' έξω πώς, ε, πού η, η πολιτική διαστρεβλώνει τα πράγματα και τον ορθολογικό συλλογισμό. Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος και έτσι πρέπει να είναι. Και πάλι υπάρχει μια ε, τάση να είναι αυτό πιο γενικό, χρειάζεται πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση στις διάφορες χώρες ούτω ώστε να εστιαζόμαστε εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Υπάρχει ανάγκη ε, να ενισχύουμε ορισμένα σώματα, ορισμένες ε, οντότητες και επιτροπές κλπ. Υπάρχουν επίσης όροι οι οποίοι βασίζονται στην απόδοση που μπορεί να αφορούν την διαχείριση δημοσίων χρημάτων, τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, της παιδείας. Αυτό εξαρτάται από τις προτεραιότητες στις διάφορες περιπτώσεις και συνήθως τα κριτήρια αυτά είναι συναφή, είναι σχετικά και χρήσιμα, αλλά δεν είναι αρκετά σαφή όπως είπα και προηγουμένως. Ε, τι είναι επίσης ικανοποιητική πρόοδος. Αυτό δεν είναι αρκετά σαφές. Υπάρχει μια ανάγκη για μια διαδικασία σαφής και ε, δομημένη για τις αξιολογήσεις και τις εκταμιεύσεις ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα έτσι όπως έχει προβλεφθεί. Ο διάλογος, ο πολιτικός σχετικά με την πολιτική είναι ένα συστατικό στοιχείο κλειδί, διότι με αυτόν τον διάλογο οι χώρες, οι δότριες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να δούνε τι αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί. Και εδώ αναφέρουμε ότι δεν έχουμε την εντύπωση ότι ο διάλογος πολιτικής χρησιμοποιείται πλήρως. Έχουμε δει παραδείγματα εκεί όπου η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εμπλακεί, όπου υπάρχει ε, πιο από μια στρατηγική πιο αποτελεσματικού διαλόγου πολιτικής και αυτό είναι ανάγκαιο. Αλλά επίσης καμιά φορά ε, δεν υπάρχει αρκετή πραγματογνωμοσύνη μέσα ε, στις διάφορες ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, ούτως ώστε να αναλάβουν αυτόν τον διάλογο πολιτικής. Το τελευταίο μου σημείο αναφέρεται στις εξωτερικές αναφορές. Είναι πολύ συχνά οι αναφορές αυτές πολύ ε, γενικές και εστιάζονται σε αυτό που δυνητικά μπορεί να βελτιωθεί και υπάρχει ε, πολύ λίγη πληροφόρηση σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο. Χρειάζεται και εδώ μια διαδικασία και αυτό απαιτεί επίσης μια μεθοδολογία αξιολόγησης. Δεν υπάρχει τέτοια μεθοδολογία τώρα. Δεν είναι εύκολο έργο βεβαίως για αυτού του είδους την βοήθεια αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα και θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε καλύτερο σύστημα αναφορών και εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα που θα έχουν επιτευχθεί. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας και τονίζοντας ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ πολύ με την γνώμη και την άποψη του εισηγητή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς ότι η στήριξη η δημοσιονομική πρέπει ή δεν πρέπει να είναι βασικός παράγον. Νομίζω ότι τα βασικά επιχειρήματα πίσω από αυτήν τη δημοσιονομική στήριξη ισχύουν ακόμα, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν για να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια καλύτερα από ό,τι επί του παρόντος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε ερωτήσεις θα είχατε να μου θέσετε. Ευχαριστώ, δίνω τον λόγο στην Επιτροπή αν θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και το ελεγκτικό συνέδριο από πλευράς μας για μια πολύ καλοσχεδιασμένη έκθεση. Ευχαριστούμε επίσης και τον εισηγητή. Είναι σημαντικό θα έλεγα αυτή η συζήτηση να τεθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν όχι μόνο σε σχέση με αυτή την έκθεση αλλά τα θέματα που αναφέρονται και στις συζητήσεις για το πράσινο βιβλίο, την το πράσινο έγγραφο το οποίο έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την <clears throat> χορήγηση απαλλαγής για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Και αυτά είναι κέρια θέματα για να υπογραμμίσουμε αυτό, να υπογραμμίσουμε την αρχή της δημοσιονομικής συνδρομής και εμείς έχουμε το μέλημα όπως και το ελεγκτικό συνέδριο να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε πείρα αρκετών ετών σε σχέση με την υλοποίηση αυτής της δημοσιονομικής συνδρομής εργαζόμαστε για αυτά τα διάφορα θέματα. Με την έγκρισή σας ο συνάδελφος Τζένκινς θα λάβει τον λόγο για να αναφερθεί εξειδικευμένα στα θέματα που προαναφέρθηκα. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όπως και ο συνάδελφο τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση και να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο για την έγκαιρη παρέμβασή τους. Έρχεται στη σωστή συγκυρία για μας γιατί όπως τόνισε ο συνάδελφος, αυτή τη στιγμή εκβάθρον αναθεωρούμε τη δημοσιονομική συνδρομή που χορηγούμε υπό το πρίσμα του πράσινου βιβλίου, του πράσινου, ε, της πράσινης ανακοίνωσης ε, που <clears throat> κατά τα τέλη του έτους ε, θα προωθηθεί. Τώρα, αρκετά από τα πολλά από τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση, θα έλεγα ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά. Αν επιτρέπετε να κάνω μόνο μία διαφοροποίηση ως παρατήρηση. Όλα αυτά θα ήταν πιο σαφή αν η έκθεση με τον ίδιο τρόπο υπεβάλλεται όπως και η ετήσια έκθεση. Θα μπορούσε αμέσως να δει κανεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παράλληλα με τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ίσως στο μέλλον μπορεί να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Υπό γενικού όρους όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειλικρινά την έκθεση την θεώρησε επικοδομητική γιατί έχει χρήσιμα, χρήσιμες παρατηρήσεις. <clears throat> Επισημαίνει τομείς που διεξοδικά θα πρέπει να εξεταστούν πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ώστε να υπάρχει ένα σαφέστερο πλαίσιο για την αξιολόγηση κινδύνων. Επίσης στο πεδίο του καθορισμού των κονδυλίων για τις επιμέρους χώρες. Επίσης ε, στον τομέα του να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο με σαφείς στόχους για τα προγράμματα και τα σχέδια αυτά. Συνδεδεμένα με όλα αυτά είναι και η ανάγκη να υπάρχει μεγάλη βελτίωση, σημαντική βελτίωση σε αφορά τον διάλογο στον οποίο θα προβαίνουμε πολιτικό διάλογο. Τούτων λεχθέντων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε πολλές περιπτώσεις ήδη προσπαθούμε να επανορθώσουμε και να θέσουμε εντάξει πολλά από αυτά τα σημεία και πρέπει να βρεθεί ο διαθρωμένος, δομημένος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Αυτό κάνουμε τώρα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία μας και τις κατευθυντήριες γραμμές ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και τις ε, κατευθύνσεις ε, του πράσινου εγγράφου. Υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε αρκετά γοργά να δράσουμε ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της δημοσιονομικής σύνδρομης. Ήδη τώρα, σήμερα, μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα όσον αφορά τους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι σαφές ότι όταν κάνει μια πληρωμή γενικής ε, συνδρομής δημοσιονομικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κάνει αυτό μετά από ε, έλεγχο και διαπίστωση ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ε, ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα. Δηλαδή, όσον αφορά το πλαίσιο, την πρόοδο, την μακρο, μακροοικονομική συνιστόσα, και ταυτόχρονα εξετάζουμε και ελέγχουμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τους δείκτες που μπορεί να συναποτελούν μέρος του προγράμματος. Έτσι θεωρούμε ότι προστατευόμαστε, αυτοπροστατευόμαστε όσον αφορά κάποιους κινδύνους. Τούτου λεχθέντος, πολλά μπορούν βέβαια να βελτιωθούν με μια πιο ενδελεχή, μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση, ώστε να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και να αντιμετωπιστούν με τα πιο εύθετα μέτρα και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, σε αυτό εργαζόμαστε. Όσον αφορά μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για τη δημοσιονομική σύνδρομη και σε συνδυασμό με την εκπόνηση της θέσης, των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν συντονισμένο διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και χωρών ε, που είναι αποδέκτες αυτής της συνδρομής. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το κατά το Συμβούλιο 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να σημειώσουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά μια πιο συντονισμένη πρόοδο στον τομέα των δημοσιονομικών και της δημοσιονομικής συνδρομής. Συνεχίζεται το έργο σε αυτό το πεδίο. Αυτό να μένετε να είναι ένα από τα στοιχεία κλειδιά που θα απορρέσουν από το πράσινο έγγραφο και ε, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις κατευθύνσεις εκείνες για να διαρθωθεί ο διάλογός μας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές ώστε να επιτευχθούν τα ευκταία αποτελέσματα των προγραμμάτων δημοσιονομικής συνδρομής από πλευράς μας. Για να επανορθώσω κάποιες παρανοήσεις που ενδεχόμενα υπάρχουν για την Γενική Δημοσιονομική Συνδρομή που παρέχεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο αυτό που έχει αναλάβει έχει αυτή την προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σωστό είναι να πει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Συνένεση από το 2006 και είναι και αυτή και η προτιμητέα μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι τριμερής η συμφωνία αυτή. Είναι τρίπλευρη. Έχει ε, συνενώσει σε μια κοινή προσέγγιση και τα τρία θεσμικά όργανα. Επίσης είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με το ποσοστό 50%. Τι έχουμε υπόψη δεσμεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μέχρι 50% της συνδρομής αυτής ε, μέσω <clears throat> κυβερνητικής ε, συνδρομής, ε, από κυβέρνηση προς κυβέρνηση. Αυτό δεν θα επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο με την γενική δημοσιονομική συνδρομή. Θα απαιτεί αυξήσεις σε τομεακή συνδρομή και σε άλλες μορφές συνδρομής που χρησιμοποιούνται μόνο εν μέρη όσον αφορά εξειδικευμένα κάποιες χώρες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό τον στόχο. Δεν έχουμε φτάσει στο 50% της ε, αρρωγής που παρέχουμε και αν συγκρίνουμε το πλαίσιο της γενικής δημοσιονομικής συνδρομής με την τομεακή εξειδικευμένη συνδρομή πόρο απέχουμε από το 50%. Μπορώ να σας δώσω μετά τη συνεδρίαση τα ακριβή μεγέθη, αριθμητικά μεγέθη. Είναι όμως σημαντικό να αποσαφινιστεί αυτό το σημείο πρώτα και κύρια. Νομίζω εδώ θα υπαρκεστώ σε σχέση με αυτό το θέμα και ολοκληρώνω. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ χρήσιμη έκθεση συνέταξε. Και εργαζόμαστε δραστήρια ώστε όλοι αυτοί οι τομείς και οι παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη μεθοδολογικά ακόμα και πριν από την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης ε, του πράσινου εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανταπόκρισης δηλαδή στο πράσινο έγγραφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα, αρχί, θα ανοίξω τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε παρακολούθησα την ε, συζήτηση την ε, πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι ικανοποιητική, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού ε, Συνεδρίου είναι τα εξής, ότι έχει κάνει η Επιτροπή σημαντικές πρόοδους, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης Υποθέτω ότι αυτή η φράση θα μπορούσε να είναι στο τέλος των περισσότερων εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχει πάντοτε περιθώριο βελτίωσης ακόμα και στην απόδοση μερικών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι, είναι τι είναι πιο αποτελεσματικό η στήριξη δημοσιονομική ή άλλη, άλλα κλασικά είδη αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν ξέρω αν είναι καλή μέθοδος αυτή η δημοσιονομική υποστήριξη. Ήμουνα το 2007 το Νοέμβριο στην Κένια ως παρατηρητής εκλογών. Ήταν μεγάλο χάος, απάτες, ε, με μεγάλη έκπληξη στις 27 Δεκεμβρίου την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους η Επιτροπή αυτόματα ε, μετέφερε 47 εκατομμύρια ευρώ στον, ε, στην, ε, στον προϋπολογισμό της Κένιας διαρθρωτική βοήθεια. Μια χώρα που εξαπατά σε μεγάλη κλίμακα όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση και άλλα. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι συστηματικά εσφαλμένο με αυτού του είδους την βοήθεια, την υποστήριξη και αφήνει ε, περιθώρια αν μερικές χώρες θέλουν να έχουν περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες μπορούν ε, να το πράξουν, διότι υπάρχουν περιθώρια, περιθώρια για πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν πάρα πολύ. Η ανάπτυξη μιας μυστικής αστυνομίας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Ποια είναι η εναλλακτική επιλογή. Εργαστικά πολύ στις, στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες, αναπτυσσόμενες χώρες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξει έλλειψη τροφίμων, ε, ε, ενέργεια, Ποια είναι η εναλλακτική λύση. άποψή μου είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια αυτά για τη γεωργία, για να έχουμε ε, είδη ρυζιού, είδη σιταριού, σίτου που να μην έχουν ασθένειες όπως επίσης και ζώα σε όλη την Αφρική. Μπορεί λοιπόν όχι μόνο ε, υπάρχει περιθώριο ε, βελτίωση, στο λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ε, το δέχομαι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα ίδια βοήθειας. Νομίζω ότι άλλες μορφές αναπτυξιακής βοήθειας για καλύτερες ποικιλίε για την γεωργία παρά να δίνουμε τα χρήματα στο γενικό προϋπολογισμό. Ο συνάδελφος Στάς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Θα έλεγα ότι είναι, μία από τις ειδικέ έκτακτες εκθέσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν και να ρίξουν φως στο τι συμβαίνει. Και χάρη στο έργο, στη δουλειά που επιτέλεσε ο Τάις Μπέρμαν και η Γραμματεία, νομίζω πολύ καλύτερα, ενδελεχέστερα μπορούμε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά της έκθεσης. Και είναι αναγκαίο και αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό υπό τους όρους του να προετοιμαστεί η χορήγηση απαλλαγής. Και αυτό είναι κάτι που πάλι αφορά και κρίσιμα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, εργάζεται από αυτού σε σχέση με το, το πράσινο βιβλίο, το ε, έγγραφο αυτό. Πραγματικά βρισκόμαστε εδώ μέσα την ζωντανή συζήτηση και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, ψηφίζοντας για την ε, έκθεση ήταν και η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για την έκθεση Γκέρενς από πλευράς της Επιτροπής Ανάπτυξης ένας ε, Λουξεμβούριος Ευρωβουλευτής ο κύριος αυτός που ασχολείται με την αναπτυξιακή βοήθεια και έχει συνειδητοποιήσει την ειδική έκτακτη αυτή έκθεση και πάλι Πρόκειται για μία από τις λίγες ειδικέ εκθέσεις που άμεσα ε, επικέντρωσε, έτυχε σε στο Ευρωκοινοβούλιο αναφερόμενη σε αυτά τα θέματα. Και αυτό κατέληξε και στην έκθεση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο γι' αυτό. Ολμάιερ παρακαλώ. Και εγώ προσθέτω τη φωνή μου στις ευχαριστίες το ελεγκτικό συνέδριο αρκετά επιχειρήματα μας έχει δώσει και μια και γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πάντα διατυπώνει με ιδιαίτερη προσοχή τις παρατηρήσεις του εγώ την έκθεση αυτή δεν την ερμηνεύω του ότι θα πρέπει η ιδιαίτερη υποστήριξη να δοθεί από το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτή τη δημοσιονομική συνδρομή, αλλά θεωρεί το ελεγκτικό συνέδριο ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν. Και γι' αυτό πρέπει με κριτικό πνεύμα να αντιμετωπίσουμε την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία άμεσα είπε ότι αυτή είναι, λέει, η προτιμητέα προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η προτιμητέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Έχω την εντύπωση ότι κάπως διαφορετικά διαπιστώνει, διατυπώνει ο Επίτροπος Πίμπαλξ στις παρατηρήσεις του από ότι η τοποθέτηση σήμερα εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή ότι πρέπει σε βάθος να εξετάζουμε και να βλέπουμε κατά πόσον η δημοσιονομική στήριξη είναι αποτελεσματική. Διότι αυτά που ανέφερε ο κύριος Μούλτερ πραγματικά λυθεύουν. Από αρκετούς συναδέφους από την ε, Επιτροπή ε, Βοήθειας για την Ανάπτυξη έχω ακούσει κριτικές παρατηρήσεις για τέτοιες χώρες όπου γίνεται λόγος για διαφθορά σε αυτές ε, και για εκείνες τις χώρες όπου έχουν αυταρχικά καθεστώτα, δικτατορικά καθεστώτα οι δικτάτορες στην εξουσία και διεφθαρμένους και κονδύλια τα οποία δεν θα πρέπει να τους ε, διατίθενται διότι τα χρησιμοποιούν για την καταπίεση και καταστολή των ιδίων των πολιτών τους και δεν θέλαμε με κανένα τρόπο δεν θέλουμε να προσφέρουμε τέτοιου είδους ε, σύνδρομη ούτε να βοηθούμε με τέτοιο τρόπο καθόλου διότι δεν ε, επαρκεί και δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της ε, η ε, χορήγηση κονδυλίων με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και η μέθοδος ε, που ακολουθείται είναι λανθασμένη. Σύμφωνα με το απόφθεγμα Πέτυχε η εγχείρηση αλλά απεβίωσε ο ασθενή. Λοιπόν, δεν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δούμε και τη στοχοθέτηση επί τη ουσία και την, να την αναθεωρήσουμε και να την προσαρμόσουμε και να επικεντρωθούμε σε τρία θέματα. Γεωργία είναι το πρώτο το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό όπω ο συνάδελφο Μούλτερ αλλά και το θέμα τη υγεία. Αν δούμε πόσο ελεηνοί είναι οι όροι και οι συνθήκε ε, στην Αφρική υπό τους οποίους όρους ε, γεννούν οι γυναίκες τα παιδιά τους εκεί οι έγκυες και πολλά από αυτά τα παιδιά πεθαίνουν τα νεογέννητα και έχουμε και θνησιμότητα μέχρι 40%. Αυτό δεν είναι επιτυχία με κανένα τρόπο και η δημοσιονομική συνδρομή δεν έχει μετριάσει, δεν έχει αντιμετωπίσει καθόλου αυτά τα προβλήματα. Και τρίτον, το θέμα της εκπαίδευσης και παιδείας και κατάρτισης. Δεν είμαι αντίθετη να δίνουμε δημοσιονομική συνδρομή και υποστήριξη, αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε έτσι στο 50% και να τα δίνουμε σε λίβδιν. Πρέπει με στοχοθέτηση, με στοχοθετημένη χρήση να διατίθενται αυτά τα κονδύλια. Είναι η καλύτερη μέθοδος αυτή έναντι άλλων κλασικών μεθόδων. Τότε μόνο είναι καλύτερα τα πράγματα. Βελτίωση ουσιαστική των πραγμάτων σε σχέση με μια χώρα. Τότε θα ήμουν υπέρ. Αν όμω είναι αμφισβητήσιμα τα πράγματα και υπάρχει, α το πω έτσι, σκιά που πλανάται για το τι συμβαίνει και όταν λένε κάποιοι, α, είναι εύκολο να τα δαπανίσει κανεί αυτά τα κανδύλια εφόσον του τα διαθέτουμε, αλλά μετά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται, δεν υπάρχει έλεγχο και αν κάτι δεν λειτουργεί καλά, ε τότε δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω λένε, ε τότε αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Μόνο όταν υπάρχει αποτέλεσμα από την βοήθεια που δίνουμε μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Αν κάτι άλλο, ένα άλλο μέσο είναι πιο αποτελεσματικό, πρέπει εκείνο να επιλέγεται. Αν ένα κράτο δεν είναι πρόθυμο να ανταποκριθεί σε εμά σε αυτή τη στοχοθέτηση, ε, θα πρέπει να επιλέξουμε τα άλλα μέσα και εργαλεία, ακόμα και αν είναι πιο περίπλοκα ή πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους. Δεν είμαι αντίθετη γενικά και ισοπεδωτικά, αλλά βλέπω τα πράγματα με ιδιαίτερα ε, κρίση, ε, κριτική ματιά, με κριτικό βλέμμα για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερα και πρέπει πολύ σοβαρά να πάρουμε το θέμα σε σχέση με την ουσιαστική στοχοθέτηση των δράσεών μας και να δούμε αν ανταποκρίνεται το σύνολο ε, του κράτους και των κρατικών πολιτικών σε αυτή τη στοχοθέτηση και να μην υιοθετούμε κάποιο άλλο γνώμονα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το σημαντικότερο συμπέρασμα νομίζω δεν το είχα σκεφτεί τόσο πολύ πριν από αυτή τη συνεδρίαση είναι η τα όσα είπε το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τον ρόλο της πολιτικής στην δημοσιονομική στήριξη. Αν χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη πολιτική μπορεί να το συζητήσουμε αυτό, αλλά τελικά χρειαζόμαστε την πολιτική. Ε, και κυρίως όταν θέλουμε να επηρεάσουμε την εξωτερική πολιτική πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ξέρουμε πού αρχίζει η πολιτική και πού τελειώνει, πού αρχίζει η πολιτική απόφαση. Ε, είναι αδύνατο να αξιολογήσουμε αν δεν ξέρουμε ε, τι είναι πολιτική απόφαση, τι είναι ουσιαστική απόφαση που βασίζεται σε άλλους παράγοντες. Κύριε Μούλντερ, είχε σημαντικό σχόλιο σχετικά με το περιθώριο βελτίωσης. Υπάρχει πάντοτε περιθώριο βελτίωσης, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι αν υπάρχει πρόοδος. Αν ε, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερο περιθώριο βελτίωσης ε, τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα θέμα ίσως ε, για το ελεγκτικό συνέδριο. Ίσως σχετικά με την διαχείριση κινδύνων. Έχουμε βελτίωση, έχουμε αντλήσει διδάγματα και τελευταίο θέμα, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, και αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Ξέρω ότι ο κύριος Χασκνένας έχει παρετηθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και θα πάει στο Ίδρυμα Νομπέλ για να εξασφαλίσει το μέλλον των βραβείων Νομπέλ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο σας, αλλά εάν θα ήθελα να του πω ότι μπορούμε τώρα να θέσουμε και ένα διαφορετικό θέμα και να ρωτήσω εάν έχετε κάποια συμβουλή. Έχουμε ε, πρώην μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου που μας έχουν πει πάρα πολλά πράγματα για τον δημοσιονομικό έλεγχο αλλά ίσως θα ήταν καλό να μας πείτε εσείς αν έχετε κανένα γενικό σχόλιο το οποίο θα θέλατε να μας υποβάλλετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μήπως έχετε κανένα γενικό σχόλιο, θα με ενδιέφερε. Ο συνάδελφος ε, Μπέρμαν για τα συμπεράσματα. Ναι, συνάδελφοι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις από όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα έλεγα πρώτα απ' όλα ε, μια γενική παρατήρηση. Αυτό το κοινοβούλιο έχει τρεις ρόλους, όπως και κάθε κοινοβούλιο. Είμαστε εδώ για να είμαστε η φωνή των ψηφοφόρων μας, είμαστε εδώ για να νομοθετούμε και είμαστε εδώ ε, για εποπτεία κοινοβουλευτική. Εάν εκπροσωπούμε τους ψηφοφόρους μας, αυτό είναι ένα ερώτημα, ένα θέμα που κάθε ευρωβουλευτής πρέπει να θέσει στον εαυτό του. Εδώ ίσως έχουμε κάποιο πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας νομοθεσία, ναι. Το κάνουμε με ενθουσιασμό, αλλά ίσως λιγότερο τους τελευταίους μήνες ψηφίζουμε πολύ περισσότερο για ψηφίσματα και όχι για νομοθετήματα. Αλλά ε, ο ρόλος μας ως εποπτικό όργανο έχει τελείως παραβλεφθεί, ίσως εκτός από αυτή την Επιτροπή. Αν έχω μόνο μερικές εβδομάδες για να συντάξω μια έκθεση για κάτι που συνεπάγεται δισεκατομμύρια χρημάτων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μπορώ να συνομιλήσω με κάποιον σοβαρά, να ερευνήσω κάτι σοβαρά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι εποπτεία παρακολούθηση κοινοβουλευτική Βεβαίω, είχα την βοήθεια του Σισκόφσκα ε, σχετικά για να εργαστώ ε, με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μερικές συνομιλίες. Γι' αυτό θα ήθελα να με συγχωρήσετε για την ποιότητα αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι το κοινοβούλιο μας χρειάζεται ενδελεχή συζήτηση για το πόσο σοβαροί θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον τρίτο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Γιάννη Μολντορ, δεν συμφωνώ γενικά ότι πρέπει να απορρίψουμε τη δημοσιονομική υποστήριξη ως μέσο. Βεβαίως και αλλού γίνονται σφάλματα. Αν δεν δεχθούμε την ιδέα ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα, τότε δεν πρέπει ποτέ να έχουμε σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες. Αν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να παίξει σχετικά με τις δυνατότητες των ανθρώπων και την ανάπτυξη ε, χωρών που δυστυχώς είχαν την κακή τύχη να είναι πτωχές, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι μπορεί και τα πράγματα να ασφάλουν ε, και θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, αλλά τα πράγματα μπορεί να μην πάνε καλά. Η συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δεν ξέρουμε πόσο πραγματικές είναι οι προθέσεις τους κλπ. Ακούσατε την έκθεσή μου ε, και είδα, είδατε πώς λέω ότι τα πράγματα πρέπει σοβαρά να αλλάξουν. Δεν πρέπει να διοχετεύουμε μόνο χρήματα, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ίδια την κυβέρνηση της χώρας και τον τρόπο που διαχειρίζεται τα κονδύλια. Ανάγκη λοιπόν να επενδύσουμε σε εποπτεία κοινοβουλευτική στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών αυτών είναι η ανάγκη να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να βοηθήσουν τους εαυτούς των. Και πρέπει να πω κύριε Μάιερ ότι ε, ότι εκεί ε, ε, ε, όπου είναι αποτελεσματική η γενική δημοσιονομική στήριξη και η τομεακή δημοσιονομική στήριξη είναι στην εκπαίδευση και στην υγεία, πληρώνοντας τους μισθούς των εκπαιδευτικών, των γιατρών, των, του νοσολευτικού προσωπικού. Γι' αυτό χρειάζεται η γενική δημοσιονομική υποστήριξη και η τομεακή δημοσιονομική υποστήριξη Γι' αυτό ζητήσαμε από το Κομισιόν 20% της αναπτυξιακής βοήθειας γενικά να διοχετεύεται προς την παιδεία και την υγεία. Και η δημοσιονομική υποστήριξη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να γίνει αυτό. Βεβαίως μπορεί να γίνουν σφάλματα, πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Συμφωνώ με τις κριτικές σας, αλλά τα παραδείγματα που επιλέξατε δεν είναι τα καλύτερα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα αν θέλετε η επιλογή είναι να χρησιμοποιούμε τη δημοσιονομική υποστήριξη μόνο αν άλλα μέσα δεν είναι αρκετά αποδοτικά και αποτελεσματικά θα έλεγα ότι ενώ η γενική δημοσιονομική υποστήριξη έχει διαφορετικούς στόχους από την υποστήριξη σχεδίων και προγραμμάτων και έργων, δεν μπορούμε να πούμε ότι αν το ένα δεν πάει καλά θα διαλέξουμε το άλλο, διότι οι στόχοι είναι τόσο διαφορετικοί ως προς την φύση τους, ώστε πρέπει να έχουμε δημοσιονική υποστήριξη για να αυξήσουμε την διαδικασία ιδιοποίησης ε, συναισθήματος ευθύνης για να βελτιώσουμε τα κοινοβούλια και πρέπει να επιλέξουμε τη γενική δημοσιονομική στήριξη αν θέλουμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές. Και μην νομίζετε ότι θα επιτύχετε κάτι σε μια χώρα όπως η Αιθιοπία ή άλλη χώρα εάν δεν έχετε γενική δημοσιονομική υποστήριξη ως μοχλό πίεση για να συνομιλήσετε με τις κυβερνήσεις αυτές σε πάρα πολλές χώρες, χρειάζεστε γενική δημοσιονομική στήριξη για να έχετε έναν δυνατό πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους ε, με τους οποίους θα δώσετε βάση στον πολιτικό διάλογο και θα ήθελα να πάρουμε σοβαρά τα πράγματα και να θεωρήσουμε ότι είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική του των λεχθέντων. Περιμένω από την Επιτροπή όλες οι κριτικές της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να ληφθούν σοβαρά υπόψη και του χρόνου να δούμε αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα στα, ε, στα σχόλια Στάς ε, Γουρμάιερ, ε, νομίζω ότι συμφωνούν γενικά με τα όσα λέμε στην εκθεσή μας. Σχετικά με τις ερωτήσεις Φέλνερ για την πρόοδο, μπορούμε να κάνουμε μια σαφή διάκριση και να δούμε ότι έχουμε διαπιστώσει πρόοδο ως προς τη διαχείριση. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε αν υπήρξε πρόοδος ως προς τη βελτίωση της χώρας. Ως προς την ουσία δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Και αυτό αναφέρθηκε από τον Ζεράρ Λοκατέλη, ο οποίος ασχολήθηκε με το λογιστικό έλεγχο. Μου είπε ότι ένας από τους λόγους που δεν προσεγγίσαμε το θέμα αυτό ρητά, το θέμα που ανέφερε ο κ. Μούλντερ, ε, αν αυτό ήταν καλύτερο από την παραδοσιακή μορφή βοήθειας είναι ότι δεν υπάρχει βάση για να κάνουμε τέτοιες αξιολογήσεις και κρίσεις. Ξέρουμε πράγματα, αλλά όχι αρκετά. Γι' αυτό υπογραμμίσαμε την ανάγκη ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για την πραγματική αξιολόγηση του τι επιτυγχάνουμε με αυτή τη βοήθεια. Θα έλεγα ότι ε, το παράδειγμα που αναφέρθηκε ε, είναι ένα παράδειγμα για το τι τα πολλά, από τα πράγματα που αναφέρουμε στην έκθεση χρειάζονται. Χρειαζόμαστε ένα καλό πλαίσιο για να κρίνουμε αν υπάρχει πρόοδος. Όπως είπε ο Κριστόβελ Φέλτνερ, χρειαζόμαστε έναν τρόπο που να μπορούμε να κρίνουμε αν η Κένια παίρνει τόσα όσα θα έπαιρνε ναι, μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε αν θέλουμε να το κάνουμε για πολιτικούς λόγους ή για τα κριτήρια που θέσατε. Και στην περίπτωση της Κένιας μπορεί να έχετε ίσως κριτήρια τα οποία θα εξαναγκάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να διοχετεύει κονδύλια. Δεν το αποκλείω αυτό. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για καλύτερη διευκρίνηση, για καλύτερα πλαίσια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η μορφή μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική όπως και άλλες μορφές βοήθειας. Σχετικά με το άλλο θέμα που ανέφερε ο Χριστόφερ Φέρερ, αν, ε, μπορώ να αναφέρω τρία μικρά σημεία, αν μου το επιτρέπει ο Πρόεδρος. Η συζήτηση η οποία προέκυψε εδώ μετά το άρθρο του Μάρτιν Βίντα εστιάστηκε κυρίως πάνω στο γεγονός ότι τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου οθούν ε, περισσότερο τις εθνικές προοπτικές παρά ασχολούνται με την προοπτικές των φορολογουμένων. Αυτά έχουν συμβεί και στο παρελθόν προτού έρθω στο ελεγκτικό συνέδριο και ακόμη και όταν ήμουν στο ελεγκτικό συνέδριο. Ήμουνα κατά οξύτατα κατά, δεν είδα τίποτα να γίνεται στα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα πράγμα. Μετά νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν μερικές σημαντικές βελτιώσεις στο ελεγκτικό συνέδριο τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να βελτιωθούν και άλλα πράγματα, αλλά έχουν βελτιωθεί μερικά. Και το σημαντικό είναι ότι είχαμε ε, βασικές αλλαγές ε, στο, στην, στην δομή μας, ε, την διοικητική Ίσως δεν έχετε δει τον αντίκτυπο. Έχουμε ε, ότι έχουμε η ευθύνη η οποία έχει κατανεμηθεί και ακόμα στους ανθρώπους που βρίσκονται στην βάση και ασχολούνται με τα πράγματα. Όχι μόνο δεν χάνουμε τόσο πολύ χρόνο σε συνεδριάσεις των 27, αλλά ακόμα πιο σημαντικό αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε υψηλότερη ποιότητα έκθεσης και ταχύτερες διαδικασίες. Επίσης τώρα έχουμε αυτό που ονομάζαμε αρχικά Management Council και μετά ονομάστηκε Administrative Committee, Διοικητική Επιτροπή, στην οποία εξουσιοδοτήσαμε για να λαμβάνει μερικές αποφάσεις. Αυτό για να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να έχουμε περισσότερη συνεκτικότητα στην διοίκηση και διαχείριση του οργάνου αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντική αλλαγή που θα έχει κάποιον σοβαρό αντίκτυπο. Ένα δεύτερο σημείο αναφέρεται στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων. Υπήρξε τάση τα τελευταία χρόνια να μετατίθενται οι πόροι εκτός από ορισμένε λειτουργίες διοικητικές και μεταφράσεις στον λογιστικό έλεγχο, στο Τα Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταφορά, η μετάθεση ήταν σημαντική. Βεβαίω, μπορεί κανείς να συζητήσει για μέρες για να μην πω για μήνες αλλά νομίζω ότι 45-50% των ατόμων στο ελεγκτικό συνέδριο εργάζονται ε, απευθείας άμεσα ε, με ε, τις, τους λογιστικούς ελέγχους. Βεβαίως ανέφερα έξοδα όπως στις μεταφράσεις στις βόρειες χώρες έχετε 60% προσωπικού που ασχολείται με λογιστικό έλεγχο. Είμαστε λοιπόν κάτω κατά 20-25% και είναι σημαντικό θέμα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στον τομέα αυτών. Και όπως είπα έχει αρχίσει η αλλαγή, αλλά πρέπει ακόμα πολύ περισσότερα να γίνουν. Θα ήθελα εγκατακλείδη να πω ότι θα μπορούσα να προσθέσω την επικοινωνία, διότι υπήρξε και εκεί κάποια βελτίωση στην επικοινωνία. Δεν θα ξοδέψω χρόνο, θα πω τελικά ότι ότι αν έχετε ένα όργανο με 27 μέλη δεν μπορείτε να έχετε πολύ αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν ε, πολιτικοί λόγοι ισχυροί για να έχει κανείς μια επιτροπή από κάθε κράτος αντιπροσωπεύεται, διότι είναι πολιτικό υλικό. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποιος από κάθε χώρα στην επιτροπή. Αυτό έχει συζητηθεί επίσης. Βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ, αλλά τα επιχειρήματα αυτά δεν ισχύουν ε, για ένα όργανο το οποίο πρέπει να κάνει κρίσεις επαγγελματικές που να βασίζονται σε σαφείς κανόνες και κριτήρια σε μια τέτοια υπηρεσία. Πρέπει να έχει κανείς μια δίκηση με 5-6 άτομα Έναν γενικό ελεγκτή, όπως έχουν πολλές χώρες, έναν γενικό... Μα δεν είναι ένα θέμα το οποίο εξαρτάται από τα μέλη. Νομίζω ότι αυτό για τα πράγματα που εξαρτώνται από τα μέλη υπάρχουν βελτιώσεις. Έχουμε ε, διαπιστώσει βελτιώσεις, αλλά για να αλλάξουμε πράγματι τα πράγματα πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στον αριθμό των ατόμων που διοικούν το όργανο αυτό που πρέπει ο αριθμός να είναι πολύ μικρότερος από ό,τι σήμερα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη και θα μπορεί έτσι η υπηρεσία να δρά με περισσότερο θάρρος και πολύ πιο γρήγορα διότι αν έχετε ένα όργανο με 27 μέλη, τότε οι αποφάσεις εξαρτώνται από τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Δεν μπορεί κανείς πάντοτε να επιτυγχάνει κονσένσους, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά από τις πολιτικές αρχές. Αυτό πρέπει να γίνει. Το οφείλουμε, οφείλουμε στους φορολογούμενους θαραλές, αποφάσεις και αλλαγές. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 12 της σημερίσιας διάταξης. Ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου διαχείριση εκ μέρου της Κομισιόν του συστήματος συνιατρικών ελέγχων επί των εισαγωγών κρεάτων μετά τη μεταρρύθμιση του 2004. Η κυρία Κιώστιγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Λαζάρου, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος του ελεγκτικού συνεδρίου για αυτά τα ε, θέματα και για την έκθεση που μας παρουσίασε αλλά και για την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε πριν ξεκινήσουμε το έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την έκθεσή της ε, σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος συνιατρικών ελέγχων επί των εισαγωγών ε, κρέατος. και που έχει να κάνει με τη διαχείριση του συστήματος των κτηνιατρικών ελέγχων μετά δηλαδή από τις ε, διατάξεις ε, για θέματα ε, υγειονομικά του 2004. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μέσα στον καμπά των ελέγχων και της τροφιμικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έρχομαι από μια γεωργική περιοχή, μια αγροτική περιοχή, τα έχετε στο έγγραφο εργασίας όλα όσα θα ήθελα να σας πω. στη σελίδα 3 έχετε τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και προς την Κομισιόν. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας αναφέρω τις τρεις συστάσεις έχουμε τη σύσταση 3 του ελεγκτικού συνεδρίου που εγώ ερμηνεύω σε εθνικό επίπεδο διότι είναι οι διάφορες εθνικές αρχές οι οποίες έχουν ένα έλλειμμα στην επικοινωνία όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η Κομισιόν θα έπρεπε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις πληροφορίες και, τη διαχείριση και την ανταλλαγή τους. Χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός. Η σύσταση 4 του ελεγκτικού συνεδρίου μιλάει για τα εθνικά σχέδια ελέγχου θα ήθελα η Κομισιόν να συμμετέχει περισσότερο και να προστατεύει περισσότερο την αρχή της επικουρικότητας και να βοηθήσει επίσης, να βοηθάει μάλλον, περισσότερο σε περίπτωση ελέγχων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο κυρίως ε, για τη χρήση ορμονών ε, ή άλλων βλαβερών ουσιών. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτούς τους ελέγχους αν η εισαγωγή κρέατος δεν επαληθεύεται και για τη διοξίνη αλλά και για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Τώρα για τις διάφορες πρωτοβουλίες ε, και νομοθετικά μέτρα που ε, ε, για τις χώρες εκείνες που δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Υποστηρίζω αυτά που προτείνει το Υποστηρίζω λοιπόν τη θέση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, και επίσης δέχομαι τους κανονισμούς, ε, θεωρώ σωστούς τους κανονισμούς 178 του 2002, 182 του 2004 Υπάρχει ένα άλλο σημείο τώρα που έχουμε στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά δεν παρουσιάζεται εδώ σύσταση είναι η ανταγωνιστικότητα των ε, ευρωπαϊκών τροφίμων έναντι εκείνων των τρίτων χωρών. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι και παραγωγοί έχουν προσαρμοστεί στις υψηλές προδιαγραφές των, ευρωπαϊκών στάνταρ. Όχι πάντα όμως αυτό ισχύει για τα άλλα προϊόντα που εισάγουμε. Όσον αφορά τώρα τις εισαγωγές για τις ζωοτροφές και ε, θέλουμε να ξέρουμε πότε θα μας απαντήσει και το ελεγκτικό η Κομισιόν σχετικά. Ο κύριος Λαζάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητήρια Ελίζαμπεθ Κόστιγκερ για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε πριν από τη συνεδρίαση ε, αυτή και διότι έλαβε υπόψη τις περισσότερες διαπιστώσεις και συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου η έλεγχη των προϊόντων κρέατος και εισαγωγών τέτοιων προϊόντων είναι μέρος της πολιτικής ασφαλείας διότι είναι σημαντικό για την ε, μετάδοση ε, νόσων ε, στους καταναλωτές. Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 4% της κατανάλωσης κρέατος και δεν υπήρξε κρίση στις εισαγωγές λόγω ελέγχου, έλλειψης, αλλά οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τους κτηνιατρικούς ελέγχους έχουν, αυξηθεί για πρόληψη και κρίζωση νόσων, έχουν ξοδευτεί πολλά ε, κονδύλια και 100 εκατομμύρια ε, για σχετικά μέτρα με την αδιατροφική ασφάλεια αλλά η κρίση διατροφική δηλαδή σχετικά με την εγκεφαλοπάθεια των οβοειδών ε, προσέθεσε σημαντικές πρόσθετες δαπάνες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτούς των κρατών μελών. Ο έλεγχος περιλήθη στο 2010 στο ελεγκτικό συνέδριο και εξέτασε την εποπτεία των, από την Κομισιόν των Κτηνιατρικών Ελέγχων στις εισαγωγές κρέατος στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που εισήχθη από τον κανονισμό 2004 που αποτελεί μέτρος, μέτρο του πακέτου υγιεινής που υιοθετήθηκε το 2006. Οι αρχές και τις συνοριακές ε, αρχές της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας και των κάτω χωρών ε, και οι έλεγχοι από, σε τρία κράτη-μέλη από την Επιτροπή Λουθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Το, οι διαδικασίες εκθήσης και ελέγχου του γραφείου εξετάστηκαν λεπτομερώς σχετικά με τον ρόλο που παίζει στον έλεγχο και παρακολούθησης από την Κομισιόν των Κτηνιατρικών Ελέγχων. Ε, μερικές οργανώσεις ενδιαφερομένων ε, ρωτήθηκαν ε, παραγωγών, καταναλωτών. Ο λογιστικός έλεγχος κατέληξε στα εξής. Η εφαρμογή της, του πακέτου Υγιεινής 2004 καθυστέρηση και πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί από ρυθμιστικής απόψεως, παραδείγματος χάρη, η ενημέρωση των συμφωνιών με τρίτες χώρες, η θέσπιση διατάξεων για ενισχυμένους ελέγχους και ενοποιημένη νομοθεσία μείωση στο επίπεδο ελέγχων εισαγωγών έγιναν δεκτές σε ορισμένες ισοδύναμες συμφωνίες με τρίτες χώρες που δεν υποστηριζόνταν από αποδείξεις δικαιολογημένες. Το σύστημα ενημέρωσης το, Traces ε, και το σύστημα έγκαιρου προειδοποίησης ε, RASF για το οποίο οι κτηνιατρικοί έλεγχοι βασίζονται, πάνω στο οποίο βασίζονται, έχουν χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ορισμένα σημεία ελέγχου συνοριακού σε τρία ε, κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιητικά και αυτό επηρεάζει την αξιοπιστία των στοιχείων και τα συστήματα πληροφοριών στο σύνολό τους. Ε, το γραφείο, η υπηρεσία αυτή εξακολουθεί να ελέγχει αδυναμίες που διαπιστώθηκαν επί τόπου ε, ε, διορθώνονται μόνο μετά από μεγάλη αναβολή. Εν κατακλείδη δείχνει ότι η κατάσταση ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καλύψουμε τις αδυναμίες. Το ελεγκτικό συνέδριο διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και να ενοποιηθεί, να ολοκληρωθεί με τρόπο φιλικό προς τους καταναλωτές, να αναπτυχθεί ε, το σύστημα, τα συστήματα Tracers και ράσφα. Ε, τρίτον, να υπάρξουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και οι δείκτες για την εφαρμογή μιας στρατηγικής για τους ελέγχους και για να προσδιοριστεί αν οι στόχοι έχουν ολοκληρωθεί να βελτιωθεί το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνων που χρησιμοποιείται και πέμπτον να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλύψουν τις αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερωτήμα. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. ευχαριστώ και σε σχέση και με το ελεγκτικό συνέδριο η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεπλάκει πλήρως στην προπαρασκευή αυτής της έκθεσης ε, σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο για την υπηρεσία που είμαι υπεύθυνο. Πάντα χαιρετίζουμε την ε, επικοδομητική τοποθέτηση του ελεγκτικού συνεδρίου και είναι χρήσιμα αυτά τα ευρήματα. Σε σχέση με τους ελέγχους έχουμε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους ε, επανειλημμένα Έχουμε απαντήσει επίσημα σε σχέση με τις συστάσεις στο ελεγκτικό συνέδριο και θα βρείτε στο παράτημα ε, συνημένα σε σχέση με την έκθεση τα στοιχεία αυτά. Σε σχέση με τα ευρήματα αυτά τα οποία πήραμε πολύ σοβαρά, όπως πάντα εξετάζουμε να δούμε πού υπάρχουν δυνατότητες για βελτιώσεις και για τομείς τόσο σημαντικούς όσο για τους ελέγχους των ζωικών προϊόντων πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Και έτσι συγκεκριμένα θα εμπλακούμε με τα κράτη-μέλη. Θα ζητηθεί από τα κράτη-μέλη η έλεγχη αυτή να προωθηθούν και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες αυτές όσο το δυνατόν πιο γόργα για να ανταποκριθούμε στις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Αν μου επιτρέπετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναφερθώ σε κάποια από τα σχόλια από την κυρία εισηγήτρια και εμείς προσβλέπουμε στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τις συστάσεις του Ελληνικού συνεδρίου και τα ευρήματά σας θα τα πάρουμε πολύ σοβαρά και προσθέτουμε ότι σε σχέση με τη δική μας υπηρεσία και τη Γενική Διεύθυνση απόλυτα θα λογοδοτήσουμε στο Κοινοβούλιο στην κανονική διαδικασία αλλά αναφέρθηκε η συγκίτρια στους ελέγχους που γίνονται στο εθνικό επίπεδο και εκεί υπάρχει έλλειμμα σε σχέση με την επικοινωνία λέγει. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφερε και το ελεγκτικό συνέδριο. Αρκετά μέτρα βρίσκονται υπό εξέλιξη για να μπορέσει το σύστημα των ζωοτροφών να βελτιωθεί και σε σχέση με τα θέματα που ευρέω αναφέρονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευρίσκονται υπό εξέλιξη αυτά και έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο κατά τα τελευταία έτη. Βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην Ολλανδία και στην Γερμανία στην εφαρμογή όσον αφορά την ιχνηλασία. Και εμεί σε σχέση με τη δική μα υπηρεσία, έχοντα πάει στην Ολλανδία και στη Γερμανία και έχοντα εξετάσει την ε, λειτουργία των ε, πραγμάτων και στι δύο περιπτώσει είδαμε σημαντικέ βελτιώσει. Θα ήθελα να προσθέσω, για να είμαστε δίκαιοι στα κράτη-μέλη που εμπλέκονται, ότι ήδη είχαν υψηλέ επιδόσει ε, από πλευρά των εθνικών συστημάτων του Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε οδήγησε στο να εγκαταληφθούν αυτά τα εθνικά συστήματα και να υιοθετηθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και σε σχέση με αυτή την προσέγγιση εμπλέκονται πλήρω ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βελτίωση τη επικοινωνία επίση και η κάλυψη αυτού του ελλείμματο. Τώρα συναντόμαστε για παράδειγμα σε τακτά διαστήματα με τι ελεγκτικέ ε, υπηρεσίε των κρατών μελών εδώ στι Βρυξέλλε ε, με πλήρη ημερήσια διάταξη των προβλημάτων που εντοπίζονται στο εθνικό επίπεδο σε σχέση με τους ελέγχους. Είχαμε επίσης ε, κατάρτιση μαθήματα σε σχέση με την βελτίωση των διαδικασιών για τα τρόφιμα και τις τροφές ε, και σε μεθοριακούς σταθμούς ε, και ελέγχους που γίνονται. Γίνονται πολλές φορές τέτοιου είδους μαθήματα κατάρτισης στα σύνορα. Αυτό σημαίνει υψηλό επίπεδο εμπλοκής στα κράτη-μέλη όσον αφορά τους ελέγχους. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο ανέφερε η συγγήτρια ήταν τα νομικά μέτρα εις βάρος των κρατών μελών, προσφυγή δηλαδή εις βάρος τους, όταν επανειλημμένα παρεκκλίνουν από το να ευθυγραμμιστούν με τις συστάσεις. Και αυτό πρέπει πολύ σοβαρά να το πάρουμε υπόψη. Είναι απαράδεκτο κράτη-μέλη επανειλημμένα να αμελούν και να περιφρονούν τις υποχρεώσεις τους. Και θα δοθεί αυστηρή συνέχεια στο θέμα. Θα ήθελα να προσθέσω όμως ότι στο θέμα των ελέγχων και της εισαγωγής ζωικών προϊόντων οι επιδόσεις είναι σχετικά καλές. Ε, γνωρίζουν και έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτών των ελέγχων τα κράτη-μέλη και τη σπουδαιότητά τους και επομίζονται με σοβαρότητα τις ευθύνες τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις, αυτό ήδη το έχουμε αναγνωρίσει και είναι δεδομένο. Επίσης αν μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε λύσεις για να ανταποκριθούμε το δυνατόν πιο γοργά και πιο αποτελεσματικά στις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Όπου είναι δυνατόν θα γίνει αυτό. Και εν τέλει, σε σχέση με την εισηγήτρια, αυτό το οποίο αφορά τις εισαγωγέ από τρίτες χώρες και σε σχέση και με το κόστος παραγωγής όταν λέει πότε μπορεί να αναμένει το Κοινοβούλιο μια έκθεση που θα καλύπτει αυτό επαρκώς. Θα ήθελα να προσθέσω ότι μόνο πολύ πρόσφατα, το Δεκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια έκθεση για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και τώρα <clears throat> βρίσκεται καθοδόν προς το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό μετά από μια πρωτοβουλία υπό τη Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δώσει και αυτό μια ευκαιρία για να έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση, όχι μόνο τέτοιου είδους συζήτηση, γιατί αναφέρεται στις ε, ασφαλέστερες εισαγωγές η έκθεση αλλά επίσης ε, να αντιμετωπίσουμε τις παρεκκλήσεις όσον αφορά και την παραγωγή και το κόστος παραγωγής σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Και πιο σημαντικό τέλος δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση τη γενική αναθεώρηση όσον αφορά τον κανονισμό για τα τρόφιμα και τι ζωοτροφέ. Υπό μία ενιαία προσέγγιση όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου θα καλύπτονται όχι μόνο για τα ζωικά προϊόντα και τα, τις ζωοτροφές αλλά γενικά και όσον αφορά ζωικά προϊόντα και τρόφιμα. Και αυτό κατά τη διάρκεια του 2012 θα υποβληθεί και θα δώσει μια πραγματική αυθεντική ευκαιρία να διεξαχθεί συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε βάθο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Ο συνάδελφο Μίλντερ. Ε, Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική έκθεση αυτή. Και είναι σκόπιμο και πρέπει να συζητηθεί σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή διότι αν έχουμε μια έκρηξη μια μολυσματική ε, ασθένεια ζώων, η επίπτωση στον προπολογισμό είναι τεράστια. Και είδαμε αρκετά παραδείγματα όσον αφορά για παράδειγμα ε, της, ε, τον αυθόδη πυρετό και την μόλυνση των χείρων και η επίπτωση στον προϋπολογισμό δημοσιονομικά είναι τεράστια. Μόνο βιαστικά φιλομέτρησα, ε, ξεφίλησα την έκθεση καθώς ε, ήρθα το απόγευμα εδώ. Είναι πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η έκθεση εξετάζει μόνο τις ε, νόμιμες εισαγωγές. Αν σε σχέση με όλα όσα πρέπει αληθεύουν στις διαδικασίες, ανταποκρίνονται στις διαδικασίες. Σε σχέση με τον αυτό διπηρετό που είχαμε πριν από κάποια χρόνια, δεν ήταν επίπτωση νόμιμων εισαγωγών, ήταν επίπτωση παράνομων εισαγωγών. Και αυτό σε σχέση με τη σύγκριση της κατάστασης στην Ευρώπη και σε σύγκριση με την κατάσταση στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία, αν περνάει κάποιος στη ΣΥΠΑ πρέπει να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο αν για παράδειγμα είχε βρεθεί σε μια τέτοια μολυσμένη περιοχή πριν από ορισμένους μήνες και έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ τα προβλήματα. Στην περίπτωση της Αυστραλίας περίπου τα ίδια συμβαίνουν όπως και εσείς είπα και εδώ σε σχέση για την α, εισαγωγή κάποιου τυριού από την Ολλανδία για συγγενείς μου, μου το πήραν από τις αποσκευές μου όταν έφτασα στην Αυστραλία. Είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη λοιπόν, ενδελεχής η έλεγχη. Αν φτάνει κανείς ε, στην Φραγκφούρτη, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους έλεγχοι επανέρχεται κάποιος από την ε, Αφρική και φέρνει τέτοιου είδους ε, πράγματα μαζί και κανένας ε, δεν το σημειώνει, δεν το παίρνει μυρωδιά. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτό συμβαίνει σε σχέση με όλους. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο πειρασμός κάποιος παράνομα να μεταφέρει κάτι από μια χώρα που επισκέφθηκε και υπάρχει τέτοιου είδους εισαγωγή από τέτοιου είδους εμπορεύματα. Πώς βλέπει το, η Επιτροπή τέτοιου είδους ε, εισαγωγές, ε, παράνομες εισαγωγές, ιδιαίτερα σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου έχουν εξαιρετικές επιδόσεις για την, ε, τον περιορισμό και αναχέτηση μολυσματικών ασθενειών. Ο Αυτόδης πυρετός ε, στην τελευταίος ε, που σημειώθηκε στη ΣΥΠΑ ήταν 1928-1930. Αυτά σε σχέση με την έκρηξη μολυσματικών ε, ζωικών ασθενειών στη ΣΥΠΑ. Εδώ έχουμε στην Ευρώπη με παράνομες εισαγωγές την, τα στοιχεία του Αυτόδου πυρετού για παράδειγμα που οφειλόταν σε παράνομες εισαγωγές για παράδειγμα από την Ινδία και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά από πλευρά της ε, ε, ιστορίας δεν έγινε χρήση της ε, επιστροφής όσον αφορά την Μεγάλη Βρετανία. Το κόστος ήταν πάρα πολύ ψηλό. Αυτό αναφέρει και η συγκίτρια σε σχέση με την έκθεσή της, το θέμα της ασφάλειας. Τι και αυτό συμβαίνει σε σχέση με την τεχνική της αντιμετώπισης τέτοιων ειδών, τέτοιων ειδών ασθενειών στην Ευρώπη. Με συγχωρείτε και το, την πολιτική σε σχέση με, την, ε, με τους εμβολιασμούς ή μη εμβολιασμούς. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Αν υπάρχει όμως μια μαζική τέτοια ασθένεια πρέπει μαζικά να θανατώνονται ζώα για να περιοριστεί η μόλυση, η, η ασθένεια στην Ολλανδία η πολιτική διαμαρτυρία θα ήταν τεράστια αν ε, συνέβαινε κάτι τέτοιο και πάλι και δεν είμαι βέβαιος αν και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν αποδεικτό κάτι τέτοιο. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια πολιτική εμβολιασμών. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας ε, δεν, ε, ε, δεν θα αποδεχόταν τέτοιου είδους προϊόντα στην Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ευρώπη, εμείς δεχόμαστε κρέας από εμβολιασμένα ζώα από τη Λατινική Αμερική και το εισάγουμε. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη ΣΥΠΑ ή με καμιά άλλη χώρα. Εμείς είμαστε εξαίρεση. Γιατί για όνομα του Θεού δεν μπορούμε να πείσουμε τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου να δέχονται αυτά τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα. Ακόμα και αν είναι για παράδειγμα το θέμα των ε, ε, γαλακτοφόρων αγελάδων. Είναι απόλυτα, θα ήταν απόλυτα ασφαλές ε, το προϊόν αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν δέχονται τέτοιου είδους αποστηρωμένο προϊόν από τέτοιου είδους αγελάδες ε, πολλές χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ η Κομισιόν για να απαντήσει στι ερωτήσει του συναδέλφου Μέλντορ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πάρα πολύ πραγματικά σκόπιμες και σημαντικές ερωτήσεις ή ε, παρατηρήσεις. Νόμιμες έναντι παράνομων ε, εισαγωγών. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Ρουμανία και ελέγχου όσον αφορά τέτοιου είδου εισαγωγέ. Όχι παραδοσιακέ εισαγωγέ σε σχέση με μεθοριακού σταθμού που είναι αντικείμενο των ε, παρατηρήσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά μεταφορέ αντικειμένων όσον αφορά ε, ταξιδιώτε σε αεροδρόμια, μέσω ταχυδρομείου, πακέτων κτλ. Δεν είναι απόλυτο το ότι αγνοούμε εμεί αυτή την υπόθεση. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να το αγνοούσαμε, όπως πολύ σωστά τονίζετε. Οι παράνομες εισαγωγές είναι πραγματική απειλή, αυθεντική απειλή. Και αν δει κανείς την πραγματική, τα πραγματικά αίτια της έκρηξης πανδημιών ή μολυσματικών ασθενειών στην Ευρώπη, οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε τέτοιου είδους παράνομες εισαγωγές. Λοιπόν, έλεγχοι υπάρχουν και γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Εσείς αναφέρατε ένα ενδιαφέρον δίλημα όταν λέτε τι γίνεται στην Ευρώπη σε σχέση με την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και σε μικρότερο βαθμό στις ΗΠΑ εδώ αντιμετωπίζουμε ε, μια μεγάλη πρόκληση σε σχέση με τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης, τον όγκο των ταξιδιωτών που μετακινούνται. Αν υιοθετούσαμε το ίδιο επίπεδο ελέγχων, υποθέτω ότι θα είχαμε μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και στα αεροδρόμια και στους μεθοριακούς σταθμούς. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα δεχόντουσαν ένα τέτοιο αυστηρό επίπεδο ελέγχων. Αυτό δεν μας αθώνει από την ανάγκη να είμαστε, δεν, δεν μας κάνει να απεμπολούμε την την ανάγκη να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε πραγματικά δραστήριοι στην εποπτεία με ελέγχου και μέσα σε ένα, από ένα διαρκή διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών δίνουμε συνέχεια στο θέμα αυτών των ελέγχων. Είναι ένα θέμα που σε σχέση με τη νέα μα έκθεση στη μεταρρύθμιση θα λαμβάνεται υπόψη που βρίσκεται υπό εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω γνωρίζει ο κ. Μούλτερ για το δεύτερο θέμα εμβολιασμοί έναντι μη εμβολιασμών. Και αυτό είναι μαζικό θέμα, ε, πολύ σημαντικό θέμα με πολύ σημαντικές διαστάσεις Υπενθυμίζω τις επιπτώσεις πριν από 10 χρόνια του αυθόδους πυρετού και των επιπτώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν θα δεχόντουσαν ποτέ πάλι να ξαναδούν τέτοιου είδους ε, ε, θανή, ε, θάνατο ζώων και την καύση τους πυρά. Όμως έχουν αναφερθεί πραγματικά εμπόδια. Πρώτον, η αποτυχία ή η άρνηση της, του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτών να δέχονται προϊόντα να καταναλών προϊόντα εμβολιασμένων ζώων. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ε, το πρόβλημα των εισαγωγών εμβολιασμένων ζώων και προϊόντων τους από τρίτες χώρες, αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται τέτοιου είδους ε, ε, αντιμετώπιση όσον αφορά μια ε, πανδημία ή μολυσματική ασθένεια. Όταν γίνονται αυτά, ε, ας το πω έτσι, μέσα στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων, αυτά μπορούν να γίνονται δεκτά. Αν όμως μέσα στο πλαίσιο μιας εκρηκτικής κατάστασης σε σχέση με εμβολιασμούς με, και έχοντας άρρωστα ζώα τα οποία αντιμετωπίζουμε, ζώα τα οποία δεν θα ήταν ε, κατάλληλα για κατανάλωση. Είναι πραγματικό αυτό το ενδεχόμενο. Ξέρουμε τι έγινε με τον αυτόδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε πολύ κοντά το Ηνωμένο Βασίλειο στο να υιοθετήσει μια τέτοια πολιτική εμβολιασμών, αλλά του είπανε οι εκπρόσωποι του λιανικού εμπορίου δεν θα μπορούμε να διοχετεύσουμε στην αγορά και να πωλήσουμε τα προϊόντα αυτά. Ένα δεύτερο, δευτερογενές θέμα είναι οι δυσκολίε για τη διαφοροποίηση προϊόντων μεταξύ εμβολιασμένων ζώων και μολυσμένων ζώων. Όπω ξέρει πολύ καλά ο κύριο Μούντερ, είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανεί από τα αντισώματα αν ένα προϊόν προέρχεται από εμβολιασμένο ζώο ή από μολυσμένο ζώο. Πρέπει να σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά την ε, επιστήμη για την διαφοροποίηση όσον αφορά τι ε, μεθόδου και τη μεθοδολογία. Είναι ένα θέμα αυτό που η κτηνιατρική κοινότητα το συζητά καθημερινά για το πώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και κάποιε εβδομάδε ε, κι κιόλα ε, στο παρελθόν είχε βρεθεί στο προσκήνιο. Θα πρέπει υπό την πολιτική υγεία ε, των ζώων, των κτηνοτρόφων, αυτά να αντιμετωπιστούν σωστά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Κιώστιγκερ για να ολοκληρώνει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ολοκληρώνοντας να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξειδικευμένη και καταλεπτόσα πληροφόρηση που μας έδωσε. Χαιρετίζουμε ότι ήδη τώρα υπάρχουν θετικές πρόοδοι που σημειώνονται. Πιστεύω ότι ακριβώς τα τελευταία θέματα που ανέφερε ο κύριος Μούλτερ καταδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι να είναι ένα ε, ασφαλές σύστημα και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με βάση αυτό. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ. Τελευταίο, σημείο 13, συγγνώμη, στην ημερήσια διάταξη παρουσίαση της έκθεσης της αντιπροσωπείας στην Ιταλία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού της 26ης ως, την 28η Οκτωβρίου του 2010. Σας έχει σταλεί σε όλους η παρουσίαση. Πρόκειται για μία αναλύση λεπτομερέστατη για όλα όσα συναντήσαμε μεταξύ 26 και 28 Οκτωβρίου στο Αμπρούτσο όπου εξετάζαμε τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων μετά από την τον καταστατικό σεισμό της Λάκουιλα και μετά η επίσκεψη στην Καμπανία όπου εξετάσαμε την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, σε ζητήματα περιβάλλοντος και για το θέμα των σκουπιδιών. Υπήρξαν προβλήματα για την χρήση των κονδυλίων αυτών στην Ιταλία. Υπάρχει το θέμα της διείσδυσης των ε, εγκληματικών οργανώσεων στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων είδαμε, διαπιστώσαμε τον κίνδυνο της διαφθοράς και ζητήσαμε ότι θα έπρεπε να αυξηθούν οι ουσιαστικοί και οι τυπικοί έλεγχοι. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία στενότερη συνεργασία μεταξύ Ιταλίας και κοινοτικών οργάνων. Την έκθεση την υποβάλαμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Αν κάποιος θέλει το λόγο για αυτό το σημείο, τότε θεωρούμε ότι εγκρίθηκε, διότι την έχουν δει και την έχουν ελέγξει όλοι οι συνάδελφοι της Επιτροπής μας. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε τη συνεδρίαση και έχουμε τώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών αν είναι παρόντες όλοι οι συνάδελφοι, αν δεν είναι θα τους τηλεφωνήσουμε.